είναι μεν αργά, αλλά η συζήτηση είχε πολύ μεγάλη σημασία για όλους και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, έτσι έκλεισε η αποψηλή μας συνεδρία. Καλό βράδυ σε όλους. Ah.